we can, manage, no problem. Mm. Dear friends, ladies and gentlemen. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ε, Ήρθε η ώρα να δούμε κάτι καινούριο στον τομέα της συνεργασίας μας, μια νέα εποχή της του δημιουργικού τομείς και τη σχετική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Πολιτισμού και της ΙΤΡΕ. Ε, Προτείναμε λοιπόν ένα νέο θέμα, τη δημιουργική βιομηχανία. Σήμερα διοργανώνουμε τη δεύτερη κοινή ε, συνεδρίαση με την Επιτροπή ΚΑΛΤ για να ανταλλάξουμε απόψεις για τις 391 ε, τροπολογίες για την έκθεση της ε, συνεκτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, τη δημιουργική βιομηχανία. Να καλωσορίσω τους ε, συναδέλφους της Επιτροπής Κάλτ και την πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Κώστα. Θα σας δώσω ενδεχομένως και τον λόγο για να μιλήσετε. Με την κυρία Κώστα θα μοιραστούμε σήμερα τις συνεδρίες και σας δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπούζεκ, με μεγάλη μου χαρά ε, συμπροεδρεύω σε αυτή τη ε, συνεδρία. Αν με επιτρέψετε να μιλήσω Ιταλικά, ήθελα να πω ότι πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την ε, πολύ σημαντική συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μας, ΙΤΡΕ και ΚΟΥΛΤ. Εδώ πρόκειται για μια στρατηγική την οποία δώσαμε ζωή κατά κάποιο τρόπο, με τρόπο ανευπροηγουμένο σε αυτή τη θητεία, μέσω ε, μια συνεργασία η οποία ξεπερνάει τα στεγανά που έχουμε συνήθως ε, εδώ στο Κοινοβούλιο για να ενδυναμώσουμε δύο πτυχές. Πρώτη, να βάλουμε περισσότερο στο επίκεντρο και να αναγνωρίσουμε περισσότερο την ευρωπαϊκή στρατηγική της Κομισιόν τα όπου μεταξύ των 10 προτεραιοτήτων δεν εμφανίζεται ο πολιτισμός, το οποίο είναι περίεργο για μια ήπειρο Ευρώπη, οπότε θέλουμε να μπει περισσότερο στο επίκεντρο όλου του Κοινοβουλίου, όχι μόνο της Επιτροπής Πολιτισμού, διότι χωρίς πλήρη αναγνώριση της αξίας του πολιτισμού, της δημιουργικότητας, ε, της ε, ε, διανοητικής ιδιοκτησίας όλων αυτών των άειλων αγαθών που παράγουν όμως τεράστια υλικά προϊόντα Χωρίς αυτά λοιπόν η Ευρώπη δεν θα έχει πολλά να πει στον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για ένα ισχυρό στοιχείο, μια στρατηγική που στοχεύει μια έξυπνη, χωρίς αποκλεισμού και βιώσιμη στρατηγική. Αλλιώς αυτά τα χαρακτηριστικά δεν θα μπορέσουμε να τα πετύχουμε. Ο δεύτερος λόγος, ξέρετε πολύ καλά ότι για μα ο πολιτισμό είναι διτό εγγενή για την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, την καινοτομία, και την αξιοποίηση και τη πολιτισμική διαφορετικότητα και τη πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά είναι και μεγάλος συντελεστής οικονομική καινοτομία, που διαδίδεται και σε άλλους τομείς και βιομηχανικός, ε, βιομηχανική συνιστόσα. Το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε στο αντικείμενο που έχουμε λάβει υπόψη για αυτήν εδώ την έκθεση ξεκινώντας από την Πράσινη Βίβλο για 12 εκατομμύρια επαγγελματίας ε, και περίπου 5 με 7% του, Ευρωπα... του ΑΕΠ ε, και 5,7% συγγνώμη του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη είναι σημαντική συνιστόσα λοιπόν αλλά έχουμε και ένα ζήτημα που αφορά τη διάσταση η κυρίαρχη διάσταση σε αυτό το τομέα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οπότε και η βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτή τη διάσταση, σε αυτά τα άλλα αγαθά και σε αυτή την αναγνώριση της δημιουργικότητας που είναι τόσο ισχυρή σε πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ακόμα και όταν δεν παράγουν πολιτιστικά αγαθά ή πολιτιστικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ πολιτιστικών επιχειρήσεων και δημιουργικών επιχειρήσεων. Εγώ πιστεύω ότι τώρα δεν έχουμε παρά να δώσουμε το λόγο, αλλά θα τον δώσει ο πρόεδρο στου συζητητέ μα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρου του Επιτρόπου Πολιτισμού τον Λουίτζι Μόργαν και όλους τους κοιόδης έκαναν εξαιρετική δουλειά. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες και ξέρω ότι ήδη διαμορφώνονται σημαντικοί συμβασμοί. Να δούμε σήμερα λοιπόν τη συζήτηση από αυτόν και όπως γνωρίζετε μετά από την ψηφοφορία που έχει προβλεφθεί για τις 9 Νοεμβρίου εμείς ε, θα μπορέσουμε, θα έχουμε δυνατότητα να ε, ε, σημειώσουμε σημαντική πρόοδο και ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιό, τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμού και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη για τη συνεργασία του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορείτε να ξαναπάρετε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, Σίλβια. Δεν νομίζω ότι θα είναι δύσκολη η συνεργασία μας γιατί συμφωνούμε επί της γενικής προσέγγισης και ξέρουμε ότι πρέπει να μοιραστούμε μεταξύ μας τις αρμοδιότητες. Οι 391 τροπολογίες είναι πολύ αριθμές, πολύ δουλειά λοιπόν για τον εισηγητή και τους συνεισηγητές και τους κεωδείς, συγγνώμη, ώστε να επιτευχθούν συμβαστικές τροπολογίες. Θέλουμε οι συμβασμοί αυτοί να είναι ολοκληρωμένοι και να συνάδουν με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε, πολύ φυσιολογικά, όπως είπε και η Σίλβια, θα δώσουμε το λόγο στους εισηγητές μας και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω τον Λουίτζι Μοργάνο, εισηγητή εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού. Έχετε το λόγο. Πέντε λεπτά ο καθένας. Και μετά, παρακαλώ συνάδελφε, έχει πάνω από τρία λεπτά για τους κοιόδη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ όλους αυτούς που συνεργάστηκαν, τους κοιόδης εννοώ, αλλά και τη γραμματεία βέβαια και τους προέδρους των δύο επιτροπών για την κοινή πολιτική βούληση. Σημαντικό να επιθυμίσουμε το ενδιαφέρον που προκάλεσε αυτή η έκθεση. Λογικό, αφού είναι κρίσιμη σημασία σε αυτές τις μηχανίες. Και για την ανάπτυξη της Ένωσης και των χωρών, αλλά και για την απασχόληση, ιδιαίτερα αυτή των νέων. Είχαμε διάφορες τροπολογίες. Θα έχουμε και τη γνωμοδότηση από την Γιούρη με καμιά πενταριά τροπολογίες που ψηφίστηκαν το πρωί. Βεβαίως, αφού ψηφίστηκαν νωρίτερα, θα τις ζούμε στη συνέχεια, όταν μας τις στείλουν. Πώς αξιολογούμε λοιπόν το θέμα των τροπολογιών. Καταρχάς, ικανοποίηση. Επειδή η μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών των συναδέλφων και ημών εισηγητών επειδή ξέρουμε ακριβώς και τον περιορισμό στο κείμενο των τροπολογιών συμπληρώνουν πλήρως το κείμενο των εκθέσεων. Πολλοί συνάδελφοι λοιπόν και από Κουλτ και από Ίντρε επιβεβαιώσαν τον πολιτικό στόχο αυτού του σχεδίου έκθεσης. Υπάρχει λοιπόν μια συνάφεια εδώ και για τους δύο και ένας κοινός στόχος. Να τροφοδοτήσουμε την Ένωση με μια βιομηχανία αυτού του είδους και κάνοντάς το αυτό να κάνουμε κάτι μακρόπνο. Η προστασία αυτών των βιομηχανιών πρέπει βέβαια να αποτελεί τμήμα και των στρατηγικών στόχων της Ένωσης σε σχέση και με το άλλο δεδομένο που γνωρίζουμε ότι το 90% αυτών των επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις με κάτω των 9 εργαζομένων μικροεπιχειρήσεις δηλαδή σε σχέση με τους απασχολουμένους. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα σε σχέση με τις τροπολογίες να υποβάλουμε και συμβαστικές προτάσεις οι οποίες θα είναι ευπαρουσιάστες και επί της ουσίας. Έχουμε στείλει στη Γραμματεία και στους Σκιώδης προτάσεις συμβιβασμών, 33 συγκεκριμένα. Λείπουν κάποιες. Το είπα και στη Γιούρη. Π.χ. copyright, δικαιώματα του δημιουργού κτλ. Στόχος κοινό και των δυο εισηγητών εδώ είναι το να καταλήξουμε σε ένα όσο πιο διαρθρωμένο κείμενο συνεκτικό και ευανάγνωστο το οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί για να ξεκινήσουμε ακριβώς πολιτικές και παρεμβάσεις όπως ζητείτε. Επί της ουσίας, δεχτήκαμε όλες τις προτάσεις που αποβλέπουν στη συμπλήρωση των αρχικών παραγράφων ας πούμε για τους στρατηγικούς στόχους στην παιδεία, κατάρτιση, επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση, στάζ, προώθηση του ευρωπαϊκού know-how, τεχνογνωσίας και άλλα θέματα που δεν θα τα παριθμίσω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεχτήκαμε επίση και αρκετά θετικά κάποιες σημαντικές πτυχές και κάναμε ομοδοποίησεις όπως οι συνθήκες των εργαζομένων σε αυτή τη μηχανία, η γενική επιχειρηματικότητα και οι προκλήσεις της ε, ψηφιακής εποχής. Υπάρχουν βέβαια κάποιες τροπολογίες που δεν μπορούμε να δεχτούμε γιατί είναι αντίθετες με την βασική πολιτική σκέψη της έκθεσης. Δηλαδή στην ουσία ζητούν την αλλαγή επί της ουσίας του αρχικού κειμένου. Έχουμε συμβαστικές προτάσεις που στάλθηκαν στους κοιόδης και στη γραμματεία. Εμείς θα θέλαμε οι συγητές να διαβουλευτούν με τις ομάδες τους και να μας στείλουν παρατηρήσεις. Από ό,τι Ξέρουμε μέχρι τις 14 του Οκτώβρη, αύριο θα πάρουμε απαντήσεις, ώστε και εμείς να αξιολογήσουμε με τη σειρά μας τις προτάσεις τους. Να δούμε αν ενδεχομένω μπορεί να υπάρξουν αντιπροτάσεις και βεβαίως στόχος μας είναι να ψηφίσουμε στις 25 Οκτώβρη στο Στρασβούργο το οριστικό κείμενο. Και ευχόμαστε να μην χρειαστούν να αλλάξουν πολλά παρά μόνο λίγες λεπτομέρειες. Συνολικά λοιπόν, θα έλεγα ότι θα περιμένω τις δικές σας παρατηρήσεις για να δούμε τι θα κάνουμε με τα θέματα που θα πρέπει να στάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Christian Eller ο συνάδελφος. Κύριε Πρόεδρε, Κώστα, κύριε Πρόεδρε, Συμφωνώ απολύτω με τα όσα είπε ο συνάδελφο. Οργάνω δεν έχω να προσθέσω πολλά. Νομίζω ότι και οι δύο οι επιτροπέ είναι ιδιαίτερω προσεκτικέ με τι ε, προτάσεις. Ε, για μας ήταν σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον να δούμε το θέμα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και πώς μπορούμε αυτό να το τονίσουμε. Αυτό που είδαμε από κοινού είναι ότι δεν πρέπει να μιλούμε μόνο για το μέλλον, αλλά και για την ε, τρέχουσα πρωτοβουλία, καθώς επίσης και για την παροχή των απαραίτητων ε, κονδυλίων για την εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπλουτίσουμε ε, τα όσα έχουμε οργανώσει και να επενδύσουμε σε αυτά που έχουμε επιτύχει. Και στο μέλλον λοιπόν ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε έχοντας υπέψη και τα ε, κονδύλια που θα τα συζητήσουμε βεβαίως και στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Συμφωνούμε λοιπόν ε, σε ό,τι αφορά την διεύρυνση ε, των ε, κονδυλίων για την Δημιουργική Ευρώπη και την διεύρυνση του και την γεφύρωση με, το, με τον ορίζοντα 2020. Και στη συζήτηση, νομίζω, στην Επιτροπή Βιομηχανία για το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να τονίσουμε την δημιουργική βιομηχανία για να, λάβουμε, να αναλάβουμε την ε, μελωδική, την ευθύνη για αυτά που μελλοντικά ζητάμε σε σχέση με αυτά που, με αυτά που θέλουμε να κάνουμε μελλοντικά, σε σχέση με αυτά που ζητούμε τώρα. Και σε σχέση με τα όσα είπε ο συνάδελφος ε, Μοργκάνο, είναι πολύ βεβαίως ε, πιο ευγενικό από μένα, από μένα Ιταλός, αλλά υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία έχουμε απορρίψει. Συνήθω υπάρχει μια τάση να υποβάλλονται ε, τροπολογίες που δεν έχουν σχέση με το θέμα της ε, ε, γνωμοδότησης, αλλά γενικώ με την ιδέα της Ευρώπης, με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτές επί της ουσίας πρέπει να τις δεχτούμε και οι δύο μεγάλες ομάδες ήδη το έχουμε κάνει. Δεν μπορώ να χρησιμοποιείτε κάθε έκθεση για να αμφισβητούμε την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό όραμα. Πουθενά δεν είναι πιο μεγάλη η αποδοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι στην, ε, στον τομέα του πολιτισμού. Εχθές, με την ομάδα ΙΝΤΑ που μελετήσαμε και από κοινού την ε, Επιτροπή ΙΝΤΑ και άλλες, Είχαμε εκπροσώπους από πολύ μεγάλες εταιρείες τη βιομηχανίας κλπ. Και σπάνια πρέπει να πω ότι η σπάνια τονίζεται όσο πολύ η Ευρώπη, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η, τα όσα έχουμε πετύχει, όσο τονίστηκαν στην α, χθεσινή διάσκεψη. Νομίζω λοιπόν ότι η, χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι ο τομέας των, της, δημιουργικής, των δημιουργικών τεχνών και του πολιτισμού είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς τομείς και κλάδους της βιομηχανίας. Και επίσης η ε, έμφαση που έδωσε και ο, ο πρόεδρος Γιούγκερ στην ομιλία του είναι αυτή που πρέπει να δίνεται στην, στον πολιτισμό. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι αυτή είναι μία από τις μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες της Ευρώπης και από την άλλη μία από, τις βασικές, από τους βασικούς ορισμούς της Ευρώπης, από τις έννοιες που ορίζουν την Ευρώπη, για το τι είναι η Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλος πολιτικός τομέας που ορίζει τόσο πολύ την ε, Ευρώπη, αλλά και που περιλαμβάνει τόσο πολλές ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον συζητητή και να ευχαριστήσω και τους δύο προέδρους που καταστήσατε ε, δυνατή αυτή την ε, συνεδρίαση και ευχαριστώ κυρίως την κυρία Κώστα γιατί μας διευκολύνει ουσιαστικά να συνεργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Είναι αρκετά καινούριος ο τρόπος αυτός ε, και να επιτυγχάνουμε τον κοινό μας ε, στόχο, ο οποίος δεν είναι κατά ανάγκη μόνο η ε, ψήφιση στην Ολομέλεια, αλλά η μετέπειτα εφαρμογή των όσων ζητούμε. Διεύρυνση λοιπόν των οικονομικών πόρων για, το, για τη Δημιουργική Ευρώπη, για τον ορίζοντα. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Έλλερ. Να ευχαριστήσω και τους δύο συναδέλφους που αποτελείται υπόδειγμα άριστης συνεργασίας και ε, ανοιχτού μυαλού του ενός προς τον άλλο. Αποτελείται υπόδειγμα. Να ζητήσω τώρα από τους κοιότητες συζητητές ε, κατά σειρά πολιτικών ομάδων να πάρουν το λόγο από ό,τι κατάλαβα από τους σοσιαλιστές έχουμε σκιώδη από την Επιτροπή Ήτρα τον Χωσέ Μπλάνκο Λόπες. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνουν τους συζητητές και να τονίσω και την αξία των τροπολογιών που εμπλουτίζουν και εμβαθύνουν την ίδια την έκθεση. Όπως και, και συμβαστικές. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τους συζητητές όπως έλεγα αλλά και τις ομάδες τους για τη θαυμάσια δουλειά τους. Μου φαίνεται ιδιαίτερα αξιόλογη και συμβαστική λύση για τους εργαζόμενους σε αυτή την βιομηχανία του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Όπως είπα στην ανταλλαγή απόψε, θεωρώ ότι αυτή η διάσταση μπορεί να συμπληρωθεί στην έκθεση εξού και οι τροπολογίες που κατέθεσα. Χαίρομαι για τις συμβαστικές προτάσεις όπου αναγνωρίζεται η ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι αυτού του κλάδου και γι' αυτό καλούμε την Κομισιόν να προτείνει λύσεις όσον αφορά την κινητικότητα εντός της Ένωσης για τους εργαζόμενους των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και να διευκολύνει και τις διαδικασίες με τρίτες χώρες ώστε να διασφαλίζονται σωστές συνθήκες εργασίας. Ζητάμε πίσω από τις χώρες μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την καλλιτεχνική δημιουργική δραστηριότητα σε σχέση δηλαδή με τις συμβάσεις, κοινωνική ασφάλιση, περίθαλψη, φορολογία τήρηση των κανόνων της Ένωσης κλπ. Και καταλήγοντας να πω ότι είναι απαραίτητο να συνδέσουμε κάποιες από συμβαστικές προτάσεις με άλλο θέμα που για μένα είναι εξίσου σημαντικό. Η σωστή αμοιβή δημιουργών και καλλιτεχνών ακριβώς για να θεσπίσουμε την προσθεμένη αξία του κλάδου αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε για τις παρατηρήσεις σας. Είσαι σκιώδης εκπροσωπούνται από τον κύριο Ευσεν Τοσενόφσκι. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους των σκιωδών εισηγητών θα του αντικαταστήσω εγώ. Ήθελα να πω κάτι για τους συναδέλφου που επισήμαναν ε, τη σπουδαιότητα της δημιουργική βιομηχανία. Ε, ίσως να είναι λίγο ομοί αυτή η ονομασία, γιατί μιλάμε για ζωντανή τέχνη. Να πω παρεμπιπτόντω ότι η μητέρα μου ήταν ζωγράφο. οπότε μεγάλωσα σε καλλιτεχνικό περιβάλλον. Αλλά η τέχνη είναι και φορέας ε, μεγάλων οικονομικών δυνατοτήτων ε, με μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι πουθενά άλλο στον κόσμο δεν είναι τόσο πλούσια αυτή η ιστορία όσο στην Ευρώπη. Οι τέχνες ε, δεν είναι απλά πνευματικές ή κάτι που μπορεί να αρέσει σε κάποιους και όχι σε άλλους. Είναι κάτι που φέρει πάνω του και πολλά οικονομικά χαρακτηριστικά και ειδικότερα για το μέλλον. Κοιτώντα τριγύρω μας, όπου και να κοιτάξουμε, όπου και να στρέψουμε το βλέμμα, υπάρχει κάπου ένα έργο κάποιο στοιχείο, design, οτιδήποτε βλέπουμε ε, διατηρεί και μεταφέρει ένα στοιχείο αυτής της παράδοσης, είναι φορέας αυτής της παράδοσης. Γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό να το ονομάζουμε πρώτα απ' όλα σωστά. Ξεκινώντας με αυτή τη σκέψη, ξεκινώντας λοιπόν από αυτή την άσχημη λέξη, τη δημιουργική βιομηχανία, τη βιομηχανία της δημιουργίας, δεν πρέπει να φοβόμαστε να παραδεχτούμε ότι οι τέχνες περιλαμβάνουν και μία οικονομική πτυχή εν γενή. Προσβλέπω λοιπόν σε μια πλήρη έκθεση που δεν έχω καμία αφιβολία θα καλύπτει όλες τις ιστορικές ε, καλλιτεχνικές πτυχές της Ευρώπης, ε, οι πτυχές αυτές που ε, συνενώνουν τα κράτη-μέλη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τωσανόφσκι. Έχουμε επίσης από την Επιτροπή μας τους σκιο, τον σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚΑ, συγγνώμη, από την Επιτροπή Πολιτισμού. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ως σκιώδης του ΕΛΚ και μέλος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μοργκάνο για τη συνεργασία που είχαμε σε αυτή την έκθεση, για την ε, συνεκτική πολιτική, για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Ε, συμφωνούμε με τις ε, τροπολογίες. Η εκπαίδευση είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα, καθώς επίσης και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Βεβαίως υπάρχει και το ότι η τροπολογία για τη συμβουλευτική για την ε, παράγραφο 9 δεν ε, έχει μπει στο κείμενο. Ε, από τη δική μας την πλευρά η κινητικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα προτιμούσαμε αυτό το τμήμα του κειμένου να ενταχθεί στο κείμενο, να παραμείνει. Ευχαριστώ. Οι περισσότεροι γεωδεις είναι απόντες. Να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο του Άλντε από την Επιτροπή Ήτρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο συγγητές για την πολύ καλή δουλειά τους σε τούτο το φάκελο. Καλωσορίζω τις ε, τροπολογίες και τις συμβολές που έχουμε λάβει για την έκθεση αυτή. Παρ' όλα αυτά, η δική μου συμβολή ε, επικεντρώνεται στις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ε, δημιουργικές βιομηχανίες στην ψηφιακή εποχή. Πρέπει να εξασχολήσουμε λοιπόν ότι θα μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή αυτή μετατροπή. Η εκπόνηση νέων επιχειρησιακών μοντέλων, πλατφορμών και καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων δίνει νέες δυνατότητες για την διάδοση του ψηφιακού περιεχομένου και νέες μορφές Αποζημίωση για τους ε, καλλιτέχνε. Επομένω, θεωρώ ότι η έκθεση αυτή επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στην ε, ψηφιακή, στην ψηφιοποίηση του ε, τομέα αυτού. Πιστεύω, όπως αναφέρεται, και από τον εισηγητή ότι οι παραδοσιακέ τα, οι συνθήκε πλαίσιο, τα προσόντα και η χρηματοδότηση φυσικά είναι εξίσου σημαντικά. Πρέπει παρόλα αυτά να επικεντρωθούμε στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξει. Όπω αναφέρεται, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές, οι, οι δημιουργικές βιομηχανίες και ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικά τμήματα της οικονομίας μας και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή των ε, παγκόσμιων αλλαγών και της καινοτομία. Πρέπει ε, να, δίσουμε, να δώσουμε στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα και, το, και τα μέσα να, ε, να καταλήξουν σε καινοτόμες ιδέες και στις εταιρείε επίση τη δυνατότητα να παραμείνουν εγκαταστημένε ή να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Επίση πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα αυτή τη έκθεση θα είναι αυτό που πρέπει. Ένα ε, σημαντικό μήνυμα ε, για να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές ε, προκλήσεις και όχι απλώς ε, μια συλλογή ευχών και επιθυμιών. Βεβαίως προσβλέπω στη συνεργασία με όλους σας έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία μου. για την ομάδα Άλντε, με εκ μέρους μάλλον Άλντε, πάμε τώρα στους πρασίνους. Έχουμε τον Μισελ Ρεϊμόν από τους πρασίνους, είναι σκιώδης από την Ήτρα και την Επιτροπή Καλτ. Η καλύτερη λύση. Σήμερα όμως αντικαθίσταται ο κύριος Ρεϊμόν από τον κύριο Μαραγκάλ από ό,τι καταλαβαίνω, που εκπροσωπεί και αυτός και δεί τις δύο επιτροπές και τους πρασίνους. Πραγματικά είστε πολύ αποδοτικός κύριε Μαραγκάλα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, δεδομένου είμαι μέλος της Επιτροπής Ήτρε και ΚΑΛΤ και αυτό μου δίνει διπλό ρόλο, ε, με διπλά πιστό σε δύο επιτροπές. Επιτρέψτε μου να περάσω ισπανικά. Ε, Δεν θέλω να υποκαταστήσω τον κύριο Ραϊμόντ. Να πω όμως κάτι το προσωπικό. Η αυτή αφορά κάτι το οποίο είναι ίδιο της Ευρώπης. Όμως, όταν μιλάμε για πολιτιστική βιομηχανία, μιλάμε για προώθηση, βοήθεια κτλ. Όταν μιλάμε αντίθετα για βιομηχανική πολιτική, μιλάμε για επενδύσεις κλπ. Αυτό που προσπαθεί να κάνει νομίζω η έκθεση αυτή είναι αυτό ακριβώς, να συνδέσει και τις δύο αυτές έννοιες ή χώρους σε πανευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο εθνικό. Νομίζω πάντως ότι αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε ότι ίσως θα χρειαστεί να ορίσουμε αυτές τις βιομηχανίες, τις πολιτιστικές και δημιουργικές. Χρειάζονται όμως παράγραφοι ολόκληρε. Κακό αυτό. Πρέπει να μην υπάρχει δυσκολία για την πρόσληψη αυτής της έννοιας, για την αντίληψή της. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε στατιστικές, δείκτες και έχουμε μία μεγάλη ποικιλία ορισμών από χώρα σε χώρα. Όταν μιλάμε λοιπόν για αυτέ τι μηχανίε, δεν εννοούμε όλοι το ίδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώ δεν θεωρώ συνετό και το λέμε σε κάποιε τροπολογίε να χρησιμοποιούμε έτσι μεγάλα στοιχεία στον ορισμό. Δηλαδή 7,5% ξέρω εγώ του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάπως περιοριστικό και δεν είναι και τόσο χρήσιμο ή σοφό. Εντάξει, να πάω στατιστικές αξιόπιστες, σωστό, αλλά τα υπόλοιπα δεν νομίζω. Μετά, χρηματοδότηση. Είναι προφανές ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν το προβλέπει αυτό. Οπότε θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τις λίγες γραμμές του προϋπολογισμού που ακριβώς αφορούν αυτές τις βιομηχανίες δημιουργία και πολιτισμού. Αλλά τέλος πάντων, επειδή ακριβώ υπάρχει δυσκολία που συνδέεται με τον προϋπολογισμό, δυσκολεύονται οι δημιουργοί να έχουν πρόσβαση ακριβώς στα διάφορα προγράμματα, κόσμε, ορίζοντας ε, 2020, Δημιουργική Ευρώπη κλπ. κλπ δεν είναι εύκολο να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Οπότε αξίζει το κόπο να στήσουμε από την Κομισιόν να αλλάξει λιγάκι τον προπολογισμό από την άποψη αυτή, ώστε να υπάρχει περισσότερη σαφήνεια. Τρίτο και τελειώνω, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση καταφτάνει ταυτόχρονα με την οδηγία για τα οπτικοακουστικά. Νομίζω θα πρέπει να απαιτήσουμε μια συνάφεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο. Αυτή η έκθεσή μας εκφράζει μια πρωτοβουλία και μια βούληση. Ίσως όμως με την οδηγία να υπάρχουν αποκλήσεις κανονιστικές. Οπότε εδώ θα πρέπει να το συνδυάσουμε. Να δούμε τι γίνεται με τις διάφορες πλατφόρμες, το ίντερνετ, ψηφιακές πλατφόρμες, πειρατεία, και πνευματικά δικαιώματα βέβαια. Θέματα πολύ σημαντικά στον κλάδο. Να πω επίσης ότι αυτός ο κλάδος χαρακτηρίζει την Ευρώπη. Καθορίζει την εικόνα της Ευρώπης και για μας αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι λοιπόν σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Γι' αυτό ακριβώς αξίζει να μιλήσουμε για προστασία για πραγματικές και ουσιώδεις ενισχύσεις προς τις βιομηχανίες αυτές που πραγματικά συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και από οικονομική σκοπιά. Να μην είναι μόνο αντικείμενο των χορηγών και το πόσο αυτή η δραστηριότητα, αλλά να τη δούμε από όλες τις πηγές της, και οικονομικές και κοινωνικές. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι που ε, ε, εκπροσωπήσατε τόσο αποτελεσματικά και τις δύο επιτροπές. Ο συνάδελφος μας ε, Κοριτσέκ από την ΚΟΕ είναι έτοιμος να κάνει το ίδιο αντικαθιστώντας τον κύριο Φερέρα και την Μαρτίνα Μιχέλης. Ο Σκιώδης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγες παρατηρήσεις θα κάνω. Ως εγώ, ως ε, προσωπικά, ως πολίτης της τσεχικής δημοκρατίας, διότι εγώ είμαι ιαλοποιός και έχω να πω ότι στο δικό μας τομέα συναντώνται η βιομηχανία και η τέχνη πολύ όμορφα και εγώ έχω ασχοληθεί και με τις μεταφορές εδώ και χρόνια δείτε όλα αυτά τα πανέμορφα κτίρια που σχετίζονται με τις μεταφορές τριγύρω μας, σύγχρονα αεροδρόμια, σιδηροδρομική σταθμή, πανέμορφα σχήματα. Όλα αυτά αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τον 19ο αιώνα όλα τα μεγάλα βιομηχανικά κτίρια είχαν κάποια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Θυμηθείτε το Bauhaus, όλες αυτές οι καθαρές γραμμές που έχουμε δει σε διάφορα κτίρια που αποτελούσαν κομμάτι του πολιτισμού μας παρότι ήταν τεράστια βιομηχανικά κτίρια. Δείτε τι δημιουργήθηκε όταν χτίζονταν οι βιομηχανίες ε, τεράστια κτίρια από τσιμέντο, όλα αυτά είναι πολιτισμός, ε, πολύ σημαντικά. Το ίδιο όταν ταξιδεύει κανείς ε, με τον αυτοκινητόδρομο από την Τσεχία μέσω Γερμανίας προς τη Γαλλία. Οι γέφυρες στην κάθε χώρα έχουν τελείως διαφορετικό σχήμα. Ε, δείτε τις γέφυρες που ε, που συνδέουν τη Δανία και τη Σουηδία, τους υπόγειους σταθμούς, τις σύραγγες. Όλα αυτά είναι βιομηχανικό design, πολιτισμός σε συγχώνευση με την βιομηχανία, όπως θα έπρεπε και στο δικό μου τομέα της αλλουργίας. Όποιο μουσείο και αν επισκεφθείτε, θα βρείτε παντός είδους ε, design σε γυαλί ε, από παλιότερες εποχές και σύγχρονα και αυτά τα αντικείμενα είναι ταυτόχρονα βιομηχανικά και αν μη τι άλλον μέρη ε, έργα Το ίδιο ισχύει και για τη βιομηχανία προσελάνης και το βιομηχανικό design διότι βρίσκεται στο όριο μεταξύ βιομηχανίας, στο σημείο επαφή μεταξύ βιομηχανίας και τεχνών και χρειάζεται λοιπόν ε, να το προστατεύσουμε. Ε, μπορεί φυσικά κανείς ε, να κατοχυρώσει κάποια αρχιτεκτονικά design. Η βιομηχανία λοιπόν ε, του πολιτισμού, η βιομηχανία και ο πολιτισμός συχνά συμβάδισαν στην Ευρώπη και συχνά στο κάθε κράτος μέλος αλλιώς γιατί είμαστε ενωμένοι στη διαφορετικότητα και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του πολιτισμού μα, ότι είμαστε ενωμένοι στη διαφορετικότητα. Γι' αυτό έρχονται τόσοι πολλοί στην Ευρώπη επισκέπτε να δουν τα κτίρια μα. Και δεν είναι απαραίτητο τα κτίρια αυτά να είναι ε, καθεδρική να ή θέατρα. Είναι και τα βιομηχανικά κτίρια, τα οποία επίση αξίζουν να απεικονίζονται σε καρτ ποστάλ. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι εξαιρετική ιδέα το να συναντηθούν δύο ε, επιτροπές μαζί και να συνεργαστούν για αυτή την έκθεση. Και είμαι βέβαιος ότι έτσι θα επισημάνουμε την ειδική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πολύ συχνά δεν αντιλαμβάνονται ούτε καν οι πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Είστε τόσο ανοιχτός που πλησιάζετε περισσότερο την Επιτροπή, τόσο την Επιτροπή ΚΑΛ, τόσο την Επιτροπή Ήτρε. Ευχαριστούμε. Έξι πολιτικές ομάδες λοιπόν, σκιώδης. Μίλησαν όλοι μόλις τώρα και οι, έξι, και οι σκιώδεις και των έξι πολιτικών ομάδων. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι της συζήτησης. Να ζητήσω από την κυρία Συμπρόεδρο, την κυρία Κώστα, να αναλάβει τα ενία της ε, συνεδρίασης. Νομίζω ότι σήμερα είχε στήσει το λόγο η Μπερές δεν ξέρω και αν από τους κοιόδες θέλουν κάποια άλλη το λόγο. Πρέπει να δώσω το λόγο βέβαια στους συζητητές και στην Κομισιόν μετά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στις επιτροπές μας που κατάφεραν να κάνουν αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι Μιλάμε για πολιτισμό, για οικονομία και για πολιτική. Και είναι αλήθεια ότι αναζητούμε χώρο δημιουργίας αξιών. Και στον τομέα του πολιτισμού έχουμε ακριβώς ένα τεράστιο δυναμικό που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί, είναι ανεκμετάλλευτο μέχρι τώρα ή όχι τελείως. Έχουμε και την παγκοσμιοποίηση η οποία αποτυγχάνει και οι πολίτες αποξενώνονται και γυρνά την πλάτη στον πολιτισμό. Η Ένωση λοιπόν δεν μπορεί μόνο να περιοριστεί στη Λευκή Βίβλο για την βιομηχανία του πολιτισμού και τη δημιουργία. Χρειάζονται συγκεκριμένε δράσει. Είπε κάποιος συνάδελφο ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την οδηγία για τα δικαιώματα των δημιουργών κτλ. Ναι, αλλά αυτό το αναφέρει και το σχέδιο μας. Αλλά έχουμε και συγκεκριμένη οπτική γωνία εμείς. Δηλαδή να εντοπίσουμε το πεδίο για το οποίο μιλάμε αυτών των βιομηχανιών. Δεν είναι και τόσο εύκολο να αποδοχτεί κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με μια βιομηχανία. Δεν είναι κάτι το κακό. Απλά και μόνο τοποθετεί στο σύγχρονο πολιτισμό, τη βιομηχανία αυτή, στο σύγχρονο κόσμο. Μετά έχουμε και το θέμα της χρηματοδότησης. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο συνδυασμό των αναγκών αυτών των βιομηχανιών χρειάζεται μια ιδιάζουσα οικονομία Γι' αυτό ακριβώς επιμένω και τονίζω την ανάγκη του ορισμού. Έχουμε μια υπερπαραγωγή χολιγουντιανή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Οπότε ο ζωγράφος ή ο φωτογράφος είναι και αυτή δημιουργοί. Οπότε όλοι αυτοί θα πρέπει να προστατεύονται από την Ένωση. Και θα ήταν άδικο και κακό να τους παρακάμψει η Ένωση. Καλό κουράγιο στους ηγητές για τη δουλειά που κάνουν. E Ευχαριστώ Νομίζω ότι δεν... χρειάζεται. Δεν έχουμε άλλε παρεμβάσεις. Να πω κι εγώ δύο πράγματα και μετά θα δώσω το λόγο στους συγγητές και μετά στην ε, Κομισιόν. Πρώτα δύο συγγητές και μετά Κομισιόν. Πρώτα Κομισιόν και μετά, αλλά τέλο πάντων. Να πω κι εγώ δύο πράγματα. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά πάνε και κάποιοι συνάδελφοι για την εμβέλεια και τη φύση των βιομηχανιών να πούμε ότι σωστά στην έκθεση γίνεται παραπομπή στην Πράσινη Βίβλο που λέει ξεκάθαρα το τι αποτελεί δημιουργία και τι πολιτισμό και οι αντίστοιχε βιομηχανίες. Είναι αυτές λοιπόν που έχουν στόχο την δημιουργία πολιστικών υπηρεσιών και η δημιουργική είναι η βιομηχανία που έχει μεγάλο περιεχόμενο δικαιωμάτων, τεχνογνωσίας, αλλά δεν είναι αυτό καθεαυτό πολιτιστικό προϊόν. Αυτή είναι η διάκριση. Το να τα θέσουμε στο ίδιο πλαίσιο δεν σημαίνει ότι τα μπερδεύουμε, απλά και μόνο προσπαθούμε να τα ενισχύσουμε. Γιατί στην πράξη αυτή η διατομιακή προσέγγιση είναι πολύ σημαντική. Εκτιμώ επίσης στα πλαίσια της άλλης έκθεσης που είχαμε που έγραψε η κυρία Έλλερ το γεγονό ότι δίνουμε σημασία και έμφαση στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο και δεν μπορεί να μας πει κάτι Κομισιόν που μόλις ξεκίνησε Ταμείο Εγγύησης, Ταμείο Επενδύσεων, που θα μπορέσει να παρέχει δάνεια, ώστε να υπάρχει ένα capability, λέει μιλήτρια, ώστε και το πιστοτικό σύστημα να προσαρμοστεί σε αυτή τη μικρότερη διάσταση την πολιτισμική και του copyright. Αλλά εμείς, όπως λέει και η έκθεση, πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη σκοπιά. Όπως έλεγε ο Μαραγκάλ προηγουμένω. Δηλαδή ζητάμε από την Κομισιόν να αρχίζει να χαράζει μια οικονομική πολιτική βιομηχανικής βάσης που θα περιλαμβάνει αυτές τι βιομηχανίες. Υπάρχει σήμερα αλλά όχι επαρκώς, αφενός και αφετέρου, να, να συνδέσουμε αυτές τις βιομηχανίες με τον ορίζοντα 2020 με το Smart Cities κλπ. Να έχουμε λοιπόν ένα πληρέστερο, ευρύτερο πλαίσιο, χωρίς να απολέσουμε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου. Αυτά. Εγώ είμαι γονή ζωγράφου και κόρη δημιουργών. Ο Γιούγκερ είχε πει ότι οι καλλιτέχνες ακριβώς είναι τα διαμάδια στο θέμα της Ευρώπης. Έχουμε την τώρα το Νίκε από την Γενική Διεύθυνση Growth και τον Κάρλο Κοράτσα, τον Γενικό Διευθυντή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της ε, Κομισιόν να παρέμβω κι εγώ. Να ευχαριστήσουμε και τους δύο εισηγητές Βεβαίω υποστηρίζουμε απόλυτα την ε, έκθεση και στηρίζουμε και την έκκλησή σας ε, για την ε, διεύρυνση των κονδυλίων για, την, για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Τώρα για τις τροπολογίες και για αυτές είμαστε σύμφωνοι. Είμαστε σύμφωνοι με τις περισσότερες προτάσεις που κάνουν οι συνεισηγητές. Να κάνω όμως κάποια σχόλια και να σας αναφέρω και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, έχουμε το πρόγραμμα Erasmus+, Έχουμε τις συμμαχίες γνώσης, όπου είναι ε, χώρος για την ε, έρευνα, για τους καλλιτέχνες, για τη βιομηχανία, να μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης υπάρχουν οι συμμαχίες προσόντων, άλλο ένα παράδειγμα, εντός του Erasmus Plus και ταυτόχρονα ξεκινούμε κάποιες ε, πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να προωθήσουν τις, ε, τα προσόντα των νέων ανθρώπων, τα επιχειρηματικά κυρίως ε, προσόντα. Να σας μιλήσω επίσης για το δίκτυο των νέων επιχειρηματιών στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, όπου προσπαθούμε να ε, δημιουργήσουμε μια ε, πλατφόρμα ε, μάθησης ομοτήμων, πρόθεσης των δημιουργών που θέλουν να γίνουν και των νέων ανθρώπων που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, σωστή δίκαιη αποζημίωση των ε, δημιουργών, ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και το γεγονό ότι δεν το έχει λάβει υπόψη στο ρυθμιστικό, το έχει λάβει υπόψη στο ρυθμιστικό πλαίσιο Κομισιόν αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το ίδιο και για το copyright, για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που ενισχύει την δημιουργία και προσφέρει κίνητρα για την καινοτομία. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία, αλλά βεβαίω συζητάτε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ναι, φυσικά η διατομιακή συνεργασία είναι σημείο κλειδί, η κινητικότητα των ε, καλλιτεχνών επίσης, γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν Είμαστε ιδιαίτερω ε, ικανοποιημένοι από την πρόταση του κυρίου Έλερ να, να, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την δημιουργική βιομηχανία. Βεβαίω, ε, σε αυτό τώρα που, λέει, που λέτε εσεί, κυρία Πρόεδρε, σε σχέση με, το, με την πρόταση που κάνετε, όταν είχαμε το 2012 ε, κάνει μια ανακοίνωση με την, για την ανάπτυξη και, την, και τις εργασίας στην Ευρώπη, τονίσαμε την δημιουργία στρατηγικών σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, ήρθαμε ε, σε επαφή με τις ε, περιφέρειες ε, σε, ένα, σε μια εκδήλωση που, εκδηλώθηκε από, που δημοργανώθηκε συγγνώμη, από την Γενική Διεύθυνση Grow για την, και για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Και αυτό που είδαμε είναι ότι οι συστάσεις από το 2012 λήφθηκαν πολύ σοβαρά υπόψη από τις περιφέρειες. Πάνω από 70 από αυτές έχουν εισαγάγει ε, βιομηχανίες δημιουργικές στις στρατηγικές τους. Και αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η στρατηγική προσέγγιση προς την καινοτομία εφαρμόζεται επί τόπου. Τέλος, και κλείνουμε αυτό, Θεωρούμε ότι η προετοιμασία για το ευρωπαϊκό ε, έτος ε, ε, πολιτιστικής κληρονομιάς το 2018 θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προσέγγιση για να προωθήσουμε τις δημιουργικές βιομηχανίες. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι μία από τις δημιουργικές βιομηχανίες ουσιαστικά. Το έτος λοιπόν θα βοηθήσει να δούμε την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο για την κοινωνία αλλά και για την οικονομία. Και εδώ ε, συνάδουμε με τα όσα είπαν και οι συναδελφοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνα και Ανάπτυξη, όπου θέλουμε να ε, επικεντρωθούμε βεβαίω και στα οικονομικά ωφέλη που μπορεί να επιφέρει ή να αποφέρει η πολιτιστική κληρονομιά. Ευχαριστούμε. Πράγματι, η πολιτιστική κληρονομιά έχει και τεράστιε προοπτικέ για αυτή τη στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κοράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως αναφερθήκε και εδώ η Κομισιόν έχει πλήρη συνείδηση της σπουδαιότητας ε, οικονομικής ε, στρατηγικής ε, των παραγωγών της βιομηχανίας δημιουργίας και του πολιτισμού. Αποτελεί και προτεραιότητα της Επιτροπής αυτής να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα τη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και έτσι, όπως είπε η συναδελφός μου, αυτή τη στιγμή μελετάμε τρεις πυλώνες. Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκότερου για τις επενδύσεις, καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για προσέλκυση βιομηχανικών επενδύσεων και την κατάρτιση στην οποία θα βασιστεί αυτός ο τομέας. Όσον αφορά το ε, ρυθμιστικό, το νομοθετικό περιβάλλον, όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή μελετάμε την αναθεώρηση της οδηγίας για την υλοποίηση ε, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την καταπολέμηση της παραποίησης. Ξέρουμε ότι η παραποίηση είναι μεγάλος εχθρός της οικονομίας μας και τροφοδοτεί τη μαύρη οικονομία και την εγκληματικότητα, το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης μελετάμε ε, προαιρετικές συμφωνίες ε, ξεκινώντα από τι ψηφιακέ πλατφόρμες. Το δεύτερο πυλόν, όπω υπενθυμίσε ο συναδελφό μου σήμερα το πρωί, μάλιστα, ε, συναντηθήκαμε με πάνω από 200 εκπροσώπους ε, κρατικών οργανισμών και βιομηχανιών για να συνεργαστούμε στο πλαίσιο τη πλατφόρμα που αναφέρθηκε πριν την Grow και την DG για τον, εξυγχρον... για τον βιομηχανικό εξυγχρονισμό. Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου Δίνουμε κίνητρα στις περιφέρειες για να αξιοποιούν καλύτερα το κοινωνικό ταμείο και τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Και επίσης και για τη δημιουργία προγραμμάτων που θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμα για τα στρατηγικά ταμεία, για τα δάνεια της Ευρωπαϊκής ε, ε, ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο τομέας της δημιουργίας και του πολιτισμού έχει να δώσει πολλά σε αυτόν τον τομέα, οπότε είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τις περιφερειές και για αυτό το σκοπό. Τέλος, όσον αφορά την κατάρτιση στην παιδεία, η Blueprint Initiative στο πλαίσιο του θεματολογίου για τις δεξιότητε έχει επιλεγεί ως προτεραιότητα. Το, επίσης η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η εκπαίδευση που σχετίζεται με τον ψηφιακό κόσμο. Όλα αυτά είναι στοιχεία κλειδιά στον τομέα των βιομηχανιών της δημιουργίας και του πολιτισμού. Ευχαριστούμε το λόγο. Τώρα έχουν οι δύο συνεισηγητές. Πρώτο ο κύριος Έλερ. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο τα όσα είπε ο κύριος Κούλιτσο και ο κύριος Μαραγάλ, για την δυνατότητα και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο Πολ Μπρακ πήγε στην ε, Γάλλος σχεδιαστής, πήγε στη Γερμανία και είχε ως ε, ε, στόχο να ασχοληθεί με την αυτοκινητοβιομηχανία να σχεδιάσει, τα, να αποτελέσει τον νέο σχεδιαστή για την αυτοκινητοβιομηχανία. Να φέρει ας πούμε την γαλλική κουλτούρα στην γερμανική τεχνική. Αλλά σήμερα 30% όλων των εσόδων της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι τα ανταλλακτικά. Γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία έχει τα δικαιώματα για, την, για το σχεδιασμό και όχι τόσο για την τεχνική. Έχει τα δικαιώματα του design για, τα, για τους καθρέφτες, ε, για, για μικρότερες αξίες ανταλλακτικά και επίσης ε, η βιομηχανία ακριβώς από αυτό τον κλάδο ε, έχει μεγαλύτερο εισόδημα από ό,τι από την κατασκευή. Και γι' αυτό αιτιολογείται και η επιτυχία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι σημαντικό λοιπόν το design. Επίσης για τις προκλήσεις. Σήμερα υπάρχουν 12 φορές περισσότερο, ε, κατεβαίνουν μάλλον από το ίντερνετ 12 φορές περισσότερο ψηφιακό περιεχόμενο από το ίντερνετ ε, σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Και αυτό έχει βεβαίως μεγάλη επίδραση ε, στις δημιουργικές βιομηχανίες. Πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι οι πλατφόρμες εισπράττουν δισεκατομμύρια και μειώνουν το, τα εισοδήματα των, δημιουργικών, των δημιουργών. τα κέρδη μένουν στις πλατφόρμες, δεν καταλήγουν στην, ε, στους α, ε, ε, δημιουργούς. Αυτό δεν είναι καλή οικονομία. Α, δεν χρειάζεται να κοιτάμε αν είναι αριστεροί δεξιοί οι, οι κυβερνώντες. το θέμα είναι της ευθύνης Εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε δεν ε, χρειάζεται να πληρώσουμε τίποτα γιατί είμαστε ε, ας πούμε ουδέτερη πλατφόρμα. Δεν γίνεται τα, οι πλατφόρμες να εισπράττουν τόσα έσοδα και να μην φτάνουν τα έσοδα αυτά ποτέ στους δημιουργούς. Έχουν, έχουμε μάλιστα 12 ε, φορές περισσότερα έσοδα για τις πλατφόρμες και μειούμενα έσοδα για τους δημιουργούς. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο δυναμικό. Και πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Δεν μιλούμε, δηλαδή, να τα κάνουμε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Δεν μιλούμε για την τεχνολογία και την τεχνική κτλ. Το θέμα είναι η δυνατότητα για τους δημιουργούς. Αλλά είδαμε πώς γίνεται, πώς φτάνουν τα κέρδη στις πλατφόρμες μεν, αλλά δεν καταλήγουν στους δημιουργούς που δημιουργούν το υλικό δε. Η ψηφιοποίηση ε, ε, θα λειτουργήσει για μας όταν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα safe harbors, τα ασφαλή, τους ασφαλείς λιμένες. Ο κύριος Μόργανο. Ο κύριος Μόργανο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια από τους σκιώδεις και λοιπούς. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για τον τομέα αυτόν. Επιτρέψτε μου όχι να απαντήσω, αλλά να επισημάνω ορισμένα πράγματα όσον αφορά τα θέματα που ακούσαμε. Πιστεύω ότι μια περίληψη για τη σημερινή συζήτηση θα ήταν η διαπίστωση του συναδέλφου Μαραγκάλ που είπε ότι η βιομηχανία της δημιουργίας και του πολιτισμού είναι το νούμερο που σήμερα χαρακτηρίζει την Ευρώπη. Μου φαίνεται μια αποτελεσματική περιγραφή σε σχέση με τα όσα ακούσαμε. Ένα δεύτερο ζήτημα. Ο Μαραγκάλ είπε ότι είναι δύσκολο σε 10 γραμμέ να καθορίσουμε τη βιομηχανία τη δημιουργία και του πολιτισμού. Αν και εγώ πιστεύω ότι πάνω από το μισό είναι η προσπάθεια να περιγράψουμε επακριβώς ε, τη συνύπαρξη όλων των πραγμάτων που αναφέρουμε μέσα. Γιατί θέλουμε να είμαστε πολύ ακριβείς διότι αν δεν αναφέρουμε ορισμένα πράγματα αυτά δεν θα ε, ληφθούν υπόψη για να χρηματοδοθούν οπότε εμείς ε, πιστεύουμε ότι έχουμε καταφέρει μια ολοκληρωμένη περιγραφή. Και μετά γίνεται και μια σημαντική προσπάθεια τεκμηρίωσης των βασικών συνιστοσών και τα δεδομένα χάρη στη δουλειά της Κομισιόν ε, επίσης. Πολλά θαυμαστά πράγματα βλέπουμε εκεί με τέτοια στοιχεία. Ε, αυτό που μας κάνει έκπληξη είναι πόσο φυσιολογικά αντιδρά ο κόσμος. Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία, θέλουμε να επιμείνουμε ως εισηγητές, διότι στην πρόταση χρηματοδότηση, εκεί όπου επανειλημμένως αναφερόμαστε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στη βούληση να γίνουν έλεγχοι των προγραμμάτων και μετά ουσιαστικά να συνδεθεί το Creative Europe, το Horizon 2020 για τα διαρθρωτικά ταμεία, ο ρόλος και οι επιπτώσεις των πολιτιστικών βιομηχανιών ώστε να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να προωθηθούν. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, για να πούμε ότι ουσιαστικά μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο, κάτι πολύ ακριβές και αυτό ακριβώς πράττει και αυτή η έκθεση. Ε, αναφέρθηκε επίσης ε, η διάσταση των οπτοακουστικών και της ψηφιοποίησης, ε, αλλά εμείς το έχουμε επισημάνει επαρκώς διότι η ψηφιακή μετάβαση είναι το στοιχείο που βοηθά τις βιομηχανίες δημιουργίας και πολιτισμού να αντικαθιστούν τις παραδοσιακές αλυσίδες παραγωγής και αξίας. Οπότε από αυτού του είδους τη σκέψη ξεκινήσαμε. Αυτό λέμε ακριβώ ε, είναι αδύνατο μια έκθεση αυτού να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ε, και φυσικά δεδομένης νέε νέες οδηγίες για τα ακουστικά θέλουμε να αποφύγουμε να υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Πιστεύω ότι συμφέρει όλους αυτό για να δοθεί εστιασμένη προσοχή και να μπορέσουμε να κινηθούμε προς την κατευθύνση που πρέπει Επίσης, η συνάδελφος Μπερέση ήταν πολύ σαφής όταν υπενθύμησε ότι πρέπει να αναφέρουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία του τομέα αυτού και τα υπόλοιπα θα τα καθορίσουμε. Και νομίζω συνέστησε μια σειρά παρεμβάσεων όσον αφορά την αμοιβή για τα δικαιώματα δημιουργού ε, εφευρέτη και τα λοιπά. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα το πρωί η Επιτροπή Γιούρη ψήφισε για τις 50 τροπολογίες και θα πάμε να δούμε και εκεί τι άλλη εγγυήση περαιτέρω δίνεται. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι επιμείναμε σε μια οδό όχι απλή, αλλά που για μας είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή πόσο είναι δυνατόν τα δικαιώματα δημιουργού να αξιολογηθούν οικονομικά. Αυτό σχετίζεται και με αυτό που ψηφίσαμε στην Ολομέλεια, στην έκθεση Κάλλας, ε, με αναφορά στις βιομηχανίες πολιτισμού και δημιουργίας. Και εκεί υπάρχει μια παραπομπή που υπενθύμησε και η Πρόεδρος για την ε, εγγύηση για την αντιμετώπιση όλων των ε, προβλημάτων σήμερα του πολιτισμού σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει μορφή όλος αυτός ο σχεδιασμός. Ε, και αυτό καθισχάζει και, μας καθισχάζει και ε, βάσει των όσων είπε η συνάδελφος ε, αυτή την ανησυχία του να προστατεύσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία με τις διάφορες πλατφόρμες που έχουμε εμφανίζονται σήμερα τους δημιουργούς και τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, ήθελα Ευχαριστώ πολύ τους συγκεκριτέ, Θα ήθελα να δώσω το λόγο, πριν δώσω το λόγο να πω δύο πράγματα. Πιστεύω ότι η συνοχή των στρατηγικών που εμείς ζητάμε με αυτή την έκθεση πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνοχή και με τις υπόλοιπες πολιτικές που αυτή τη στιγμή εξετάζονται στις διάφορες επιτροπές. Σκέφτομαι τις διάφορες οδηγίες για το copyright, τα ζητήματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να υπάρχει συνοχή, ε, να αναγνωρίζεται η κεντρική αξία των δημιουργών και της δημιουργικότητας ως βασικού στοιχείου της αλυσίδας αξιών και οι ίσες συνθήκες ανταγωνισμού που πρέπει να διασφαλίζονται επειδή υπάρχουν χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και καθηκόντων και υποχρεώσεων όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Μόργανο. Για να κλείσω όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τα διαδικαστικά. Έτσι όπως συμφωνήθηκαν, συνάντηση των σκιωδών ανακοινώθηκε πριν από λίγο για να επιληθούν τα εκκρεμή ζητήματα για τα συμβαστικέ τροπολογίε. Ξέρουμε ότι ακόμα έρχονται προτάσει από την ε, Γιούρι, 25 ε, Οκτωβρίου στο Στρασβούργο θα στείλει γραμματεία μια λίστα ψηφοφορία και ε, ξεχωριστά σχόλια για τα διάφορα τμήματα με προθεσμία 7 Νοεμβρίου ώστε η τελική λίστα ψηφοφορία να μπορεί να σταλεί έγκαιρα για την ψηφοφορία που θα λάβει χώρα στην Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου. Αυτά τα είναι τα διαδικαστικά. Να ξαναευχαριστήσω όλους για την παρουσία τους, στην Κομισιόν, τις δύο γραμματείες των Επιτροπών μας και φυσικά την ευγενική ε, συνεργασία του Προέδρου Μπούζεκ. Ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά συναρπαστική συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστήσω ε, και την κυρία Μπέρες, πραγματικά ήταν συναρπαστική συζήτηση. Κυρία Μπέρες, ε, κινητή υγεία σε 10 λεπτά. M-Health γιατί η υγεία καμιά φορά είναι πιο σημαντική από τον πολιτισμό. Λυπάμαι που το λέω. Φεύγει όμως η κυρία Μπέρες. Ε, γνωμοδότηση της Γιούρη ε, ψηφίστηκε και θα πάει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας. Επόμενη συνεδρίαση την 5η 10 Νοεμβρίου. 10 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες εδώ. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για τη συνεργαστική συζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι από την Ήτρε, αλλά και από την Κούλταν θέλετε να μείνετε, είσαστε πολύ ευπρόσδεκτοι. M-Health. Και εδώ από κοινού η, η ακρόασή μας με την Επιτροπή ΕΜΒΗ. Σε 10 λεπτά, όχι μεγάλο διάλειμμα, μην απομακρυνθείτε.